Περνάμε λοιπόν στην ε, ε, έκθεση από την πλευρά του συναδέλφου Σμιθ ε, σε ό,τι αφορά το Χονγκ Κόνγκ 20 χρόνια μετά την παράδοσή του. Οπότε δίνω κατευθείαν το λόγο στον συνάδελφο για να κάνει την παρουσίαση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομη θα είναι η παρουσίασή μου, πράγμα νομίζω πως θα σας χαροποιήσει. Ε, εδώ θεωρώ ότι έχουμε να κάνουμε ένα ζήτημα όπου έχει προστιθέμενη αξία Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συμβάλλει εδώ ε, επικοδομητικά. Νομίζω πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε τους ιστορικούς ε, δεσμούς των κρατών μελών μας έτσι ώστε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για την άσκηση της εξωτερικής μας πολιτικής ανά τον κόσμο. Δηλαδή να μπορούμε να ασκούμε την πολιτική μας χωρίς να είμαστε είμαστε όμοιροι των ιστορικών γεγονότων. Ε, ωστόσο, ε, ε, αποτελεί τραγωδία για μένα το γεγονός ότι καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να μιλάει με μια ενιαία αφωνή, η δική μου χώρα αποφάσισε να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρότι η Σκοτία, η δική μου ιδιαίτερη ε, πατρίδα θα συνεχίσει τους στενούς της δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση στο Χονγκ 20 χρόνια μετά από την παράδοσή του από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Κίνα και στο πλαίσιο τη δέσμευση που ανέλαβε και εκείνα για αυτά τα 50 επόμενα χρόνια. Αποτελεί βέβαια σημαντικό εμπορικό εταίρο ε, το ε, αλλά και σημαντικότερο στο πλαίσιο του διαλόγου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Και παρότι είναι πραγματικά ένα ε, εντυπωσιακό μέρος ε, το Hong Kong, υπάρχουν προβλήματα και πράγματι έχουμε την αίσθηση ότι υπονομεύεται το σύστημα των δύο συστημάτων μίας χώρας όπως αναφέρουμε ειδικότερα στα σημεία B και L. Ε, υποστηρίζουμε επίση, στην παράγραφο για παράδειγμα 5, ότι θα πρέπει να την χάνει η ελευθερία τη έκφραση. Επίση, στην παράγραφο T αναφερόμαστε στου τρόπου με του οποίου μπορούμε να υποστηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών εντό του Χονγκ Κονγκ, ειδικότερα κάποιε ομάδε ε, των οποίων το έργο δυσχεραίνεται όλο ένα και περισσότερο. Ε, επιχαίρω το γεγονό ότι έχουμε φτάσει σε ε, μεγάλο βαθμό ομοφωνία ε, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μόνο δύο τροπολογίε από την πλευρά τη GUNGL ω προ τι περισσότερε προσπάθειε που θα πρέπει να γίνονται για την καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και του ξεπλήματο χρήματο. Πράγματι πρόκειται για σημαντικού τομεί και του υποστηρίζουμε και εμεί. Θα πρέπει να ενταθεί η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό τον των ε, Πρασίνων, δηλαδή ε, την γραμματεία του, του Κοινοβουλίου και όλου του συναδέλφου για την ε, συνεργασία μα. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Επίτροπο Άντριου Κάτη για να μα εκφράσει τη σκέψη του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το Hong Kong είναι ο, ένας πολύ σημαντικός εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, πάνω από 2.000 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ε, έχουν παρουσία στο Χονγκ Κονγκ και η Ευρώπη είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ε, εμπορικός εταίρος του Χονγκ Κονγκ μετά την Κίνα. καλέσαμε τους εκπροσώπους του Χονγκ να μας ε, επισκεφθούν στις Βρυξέλλες το συντομότερο. Και ε, η αυτονομία του Χονγκ θεωρούμε ότι ήταν η βάση για την επιτυχία. Οι πολίτες ε, θέλουν να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις και να γίνουν εκλογές για το νομοθετικό και εκτελεστικό συμβούλιο αλλά βεβαίως η αρχή μία χώρα, δύο συστήματα ε, έχει, δέχεται συνεχείς πιέσεις. Το κράτος δικαίου και η ανεξαρτησία της ε, δικαιοσύνης στο Χονγκ Κόνγκ έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση. Η μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας έχει αναβληθεί. Ε, ε, και δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε την περίπτωση πέντε εκδοτών οι οποίοι εξαφανίστηκαν, απήχθησαν το 2015. Αυτή ήταν μια τεράστια ε, πρόκληση, για ε, τεράστια παραβίαση κατά τη δική μας άποψη. Στη συμφωνία με την έκθεση θέλουμε να ανισχύσουμε τη διμερή συνεργασία με το Hong Kong ο τελευταίος διαφερμένος διάλογος με το Χονγκ Κόνγκ έλαβε χώρα λιγότερο πριν από ένα μήνα. Η βασική αρχή, μια χώρα, δύο συστήματα, θεωρούμε ότι είναι ουσιαστική για την ευημερία του Χονγκ Κόνγκ. Ε, ωστόσο υπάρχει το πρόβλημα με την Κίνα οι δικές μας σχέσεις με την Κίνα εντατικοποιούνται όχι μόνο όσον αφορά το, τις εμπορικές ανταλλαγές αλλά και, τα, και άλλα θέματα εξωτερικής ε, πολιτικής. Ε, θεωρούμε ότι η διαφύλαξη της αρχής μιας νέας χώρας είναι υπέρ του συμφέροντος και της Κίνας. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σουίτσα έχει το λόγο εκ μέρους του ΕΛ και 1,5 λεπτό. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την συνεργασία και την αμοιβαία υποστήριξη που είχαμε είναι μια σύσταση προς την Επιτροπή, το Συμβούλιο και την ε, είπατε εκπρόσωπο. Γι' αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι στην έκθεσή μας είπαμε ότι το Hong Kong είναι σημαντικός εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως υποστηρίζουμε τόνο την ε, προσέγγιση μία χώρα, δύο συστήματα, ε, καθώς και τον υψηλό βαθμό αυτονομίας που έχει το Hong Kong σε σύγκριση με την Κίνα. Γι' αυτό και αυτό διατυπώθηκε και στην κοινοβρετανική διατήρηξη πριν από 20 χρόνια. Ε, εμείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχουμε υποστήριξη προς όλους τους εμπορικούς μας εταίρους. Γνωρίζουμε ότι στο Χονγκ Κόνγκ ε, υφίσταται το κράτος δικαίου και υπάρχει εγγύηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλουμε μέσω της έκθεσης αυτής να υποστηρίξουμε περαιτέρω τους πολίτες του Χονγκ γιατί ο στόχος μας είναι να γίνει πιο φιλελεύθερη και η κινέζικη, η κινέζικη κοινωνία ε, και το Χονγκ εδώ μπορεί να είναι ένα εργαλείο. Όσον αφορά τις εκλογές, οι προσεχείς εκλογές θα πρέπει να είναι απολύτως δημοκρατικές και διαφανείς, αλλά βεβαίως θα πρέπει να ενισχυθεί και ο διμερής ε, διάλογος και αυτό το τονίσαμε ε, μέσω της ψηφοφορίας που έγινε στην ΑΦΕΤ. Τώρα έχει το λόγο ο κύριος Πίτσουλα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αντιπρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια ε, για την έκθεση αυτή. Είναι σημαντικό βήμα για την περαιτέρω συνεργασία με το Hong Kong. Έχουμε 20 χρόνια πίσω μας, 30 χρόνια έχουμε μπροστά μας. Η βασική αρχή ε, μία χώρα, δύο συστήματα είναι σημαντική. Θα πρέπει να υπάρχει βελτίωση της συνεργασίας όσον αφορά τα εκπαιδευτικά προγράμματα, παραδείγματι. Τώρα, όσον αφορά την κατάσταση στο Hong Kong, ε, διαπιστώνουμε την παρέμβαση του Πεκίνου ε, στο Χονγκ Κόνγκ, για παράδειγμα η προσπάθεια ρίχνωση των ελευθεριών των δημοσιογράφων. Ε, ωστόσο, η επίσημη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια νέα Κίνα, δύο συστήματα. Γι' αυτό θα ήθελα, και θα ήθελα επίσης να επισημάνω ένα περαιτέρω πρόβλημα, την φοροαποφυγή και φοροαπάτη και θα ήθελα να απευθύνω έκκληση προς την κυβέρνηση του Χονγκ Κόνγκ να λάβει μέτρα κατά επιχειρήσεων που ε, καθιστούν δυνατές τέτοιου είδους ε, καταχρηστικές ε, πρακτικές. Ο κύριος Μπέλτερ έχει το λόγο. Ε, στο New York Review of Books διάβασα ε, στο τελευταίο τεύχος ε, ένα άρθρο σε σχέση με τις διαμαρτυρίες στο Χονγκ Κόνγκ Εκεί λοιπόν αναφέρθηκαν μία σειρά από υπερασπιστές ε, των βασικών δημοκρατικών αξιών, οι οποίοι όλοι τους το σύνολό τους ε, ουσιαστικά αναφέρθηκαν στην υπονόμευση αυτού του συστήματος ε, μίας χώρας δύο συστημάτων, ουσιαστικά δηλαδή αυτού του πλουραλιστικού συστήματος στην Κίνα. Αυτό λοιπόν πολύ σωστά αναφέρει και ως βασικό σημείο έκθεση του συναδέλφου δηλαδή, ε, πραγματικά θα ήθελα να γίνει μια περαιτέρω συζήτηση σε σχέση με αυτήν την ε, έκθεση, γιατί πραγματικά μια τέτοια έκθεση μπορεί να δώσει περισσότερη δύναμη σε αυτούς τους υπερασπιστές ε, της δημοκρατίας στο Χονγκ Ευχαριστώ. Λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Σέντοβαν έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω πως ε, θα πρέπει να διατηρήσουμε ένα ανοιχτό πνεύμα όταν προσεγγίζουμε αυτό το ε, αφιλογόμενο ζήτημα της ε, Κίνα. Από τη μία πλευρά έχουμε την υπονόμευση αυτού του συστήματος μία χωρα δύο συστημάτων, αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να ασκήσουμε κριτική και στην ε, πολιτική που έχουν ασκήσει διάφορε ελίτ ε, στο Χονγκ Κόνγκ και η οποία έχει οδηγήσει σε μια ισχυρά πολλωμένη κοινωνία που έχουμε δηλαδή ένα τμήμα τη κοινωνία που είναι πάρα πολύ εύπορο και ένα άλλο τμήμα το οποίο ζει σε ακραία ε, πραγματικά οι, τα ε, μέσα ενημέρωσης έχουν αναφερθεί σε κρίση η οποία έχει προκύψει τα τελευταία ε, χρόνια ε, ε, και η οποία έχει προκύψει και από διάφορα χρήματα τα οποία δεν έχουν προέρθει από νόμιμες δραστηριότητες και δεν αναφέρονται ως τέτοια, δεν δηλώνονται ως τέτοια. Οπότε δεν ξέρουμε ε, πώ μπορούμε να αναφερόμαστε σε έναν αξιόπιστο εταίρο υπό τέτοιε συνθήκε και εμεί από την πλευρά τη δική μα πολιτική ομάδα δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε κατά συνέπεια αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Ε, λέει η Πρόεδρος ε, και εκ μέρους της ε, Επιτροπής και πάλι ο Επίτροπος Αντριουκάτης έχει το λόγο. Η διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑ δεν θα τηρηθεί λόγω της του χρόνου. Πολύ σύντομη αυτή η ανταλλαγή απόψε και εκ μέρους Αντιπροέδρου της Φεντερίκα Μογκερίνη θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή έξοχη δουλειά του ευχαριστώ και τα μέλη για αυτά που είπαν συμπεραίνουμε τη συζήτηση ότι όλοι έχουμε κοινό στόχο την υποστήριξη αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ και, ότι, και της αρχής μια χώρα δύο συστήματα. Οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσης και Χονγκ Κονγκ ε, βελτιώνονται. Δεν αφορούν μόνο εμπόριο και οικονομικά θέματα, αλλά τελωνιακή συνεργασία, καινοτομία, τεχνολογία, ανταγωνισμό, ασφάλεια τροφίμων, περιβάλλον, εκπαίδευση. Οι εταιρείε Ευρωπαϊκή Ενώσεω παίζουν σημαντικό ρόλο στην παροχή χρηματοστατικών υπηρεσιών, στο λιανικό εμπόριο, μεταφορές, επιμελητεία. Όλα είναι ζωτική σημασία για το Χονγκ Κόνγκ. Υπάρχει επιχειρηματικό περιβάλλον αποτελεσματικό στο Χονγκ Κόνγκ και ελπίζουμε ότι θα διατηρήσει τα υψηλά πρότυπα στον φωτοκράτο δικαίου, τη διαφάνεια, μη διάκριση και οικονομική ελευθερία, ότι θα διατηρηθούν και στο μέλλον. Κλείνοντα, να επισημάνω εκ νέου ότι εκτιμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ρόλο του Κοινοβουλίου που διατηρεί στο διεθνέ θεματολόγιο, στη διεθνή ατζέντα αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Ανδρουκάητη. Και κλείνοντας, δίνω το λόγο στον συγκητή. Πάμε σύντομο, συμφωνούμε με τι εκθέσεις, έγινε η δουλειά. Πριν φτάσουμε στην Ολομέλεια, προσβλέπω σε υποστήριξη από την πλειοψηφία αύριο πράγματι όσον αφορά τον εκλογικό νόμο και τη μετανάστευση αυτού στο σημείο H το καλύπτουμε αυτό ε, και είναι ισορροπημένο το κείμενο. Ευχαριστώ τους συναδέλφους πάρα πολύ καλή δουλειά και προσβλέπω στην αυρινή ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Ε, υπέροχα λέει πρόεδρος. And we are